Ε, buongiorno Χαίρετε. Να ξεκινήσουμε τη συνέδρια της Επιτροπής Γυναικών. Σήμερα θα προεδρεύσω εγώ, αντικοθεστώντας ε, την Πρόεδρο και τις πρώτες αντιπροέδρου. Θα ξεκινήσουμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν ε, στάσεις μπορούμε να την εγκρίνουμε. Αύριο θα προσθέσουμε στην ημερήσια διάταξη μετά από το σημείο 14 ψηφοφορία για τις ε, τροπολογίες ε, για το Gender Mainstream έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, της συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για τη δημοκρατία και τα κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης ε, της 17ης και 18ης Φεβρουαρίου της Επιτροπής. Αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσεις εγκρίνουμε και τα πρακτικά. Σημείο 3. È possibile inviare proposte per nuovi progetti. Μπορείτε να στείλετε προτάσει για νέα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικές δράσει ή προτάσει για παράταση ε, των πιλωτικών προγραμμάτων για το 2017. Η προθεσμία είναι 29 Απριλίου, 12 το μεσημέρι. Για την υποβολή των τροπολογιών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ε, διαθέσιμη πλατφόρμα που έχουμε στο e-committee. Και περνάμε τώρα στο σημείο 4. το οποίο θα το εξετάσουμε μαζί με το σημείο 5 διότι πρόκειται για δύο εκθέσεις οι οποίες ε, είναι αλληλένδετες. Το ένα είναι η εφαρμογή του άλλου. Έχουμε την έκθεση για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγήτρια είναι η κυρία Κατρίν Μπαρτέρ, στην οποία δίνω και το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ. να σχολιάσω πρώτα απ' όλα αυτή την έκθεση για την εμπορία ανθρώπων σε εξωτερικέ σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την επόμενη. Λοιπόν, εμπορία ανθρώπων από τρόπεο ε, ε, έγκλημα ε, σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πραγματικά συμβαίνει παντού. Όπου και να μένετε στην Ευρώπη θα είσαστε σίγουρα κοντά σε μια περίπτωση ε, ε, ελεγχόμενων ανθρώπων που ζουν σε κατάσταση δουλείας ε, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας. Έχω κάνει 62 πολλά χρόνια αυτό το ζήτημα και χαίρομαι που το ανέλαβα εδώ στο Κοινοβούλιο. Ελπίζω να βοηθήσω με, με αυτήν για την καταπολέμηση, με αυτή την έκθεση για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Ευχαριστώ τη Γραμματεία της Επιτροπής, ε, τη σύμβουλό μου, αλλά και τους ε, συναδέλφους ε, και τους υπαλλήλους της Επιτροπής που με βοήθησαν. Ήταν αγαστή συνεργασία με τους συνεισηγητές Λόχ Πίλερ και Βαλέρα. Ε, υπάγεται στο άρθρο 54 η έκθεση και είναι τρεις οι συναρμόδιες επιτροπές, είναι λίγο περίπλοκη, περίπλοκη διαδικασία. Η, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων η κυρία Λόχπιλε έχει ένα ξεκάθαρο μια ξεκάθαρη άποψη σε σχέση με τις αρμοδιότητες σε κάθε συναρμόδιας επιτροπής, οπότε μας βοήθησε εμένα και την κυρία Βαλέρα να ξέρουμε τι υπάγεται σε αρμοδιότητες ποιας επιτροπής. Ε, και έτσι έγινε η κατανομή αρμοδιοτήτων ανάμεσα στις τρεις επιτροπές. Ε, το σημαντικό για μένα είναι να αποδοθεί έμφαση στη διάσταση των δύο φύλων για την καταπολέμηση του φαινομένου εμπορίας ανθρώπων στις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στην έκθεση Επιτροπής Γυναικών. Είχαμε αυτό το περιορισμό για τον αριθμό χαρακτήρων. Παρ' όλα αυτά, έβαλα τα δυνατά μου για να καλύψω όλα τα βασικά ζητήματα. Παραδείγματο χάρη, ανθρώπινη προσέγγιση για την καταπολέμηση αυτή τη αξιόπινη πράξη και εγγραφή του ε, τη καταπολέμηση σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Κοινωνικέ ανισότητε, όπω τονίζω, ε, εντείνουν το φαινόμενο και αυτό εντείνεται επίση και από τα θέματα σεξουαλική βία και διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών. Ε, η ΔΕΛΤΑ Ανάπτυξη και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση ε, καλούνται στι εξωτερικέ σχέσει να προσφέρουν ε, καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίε που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση των δύο φύλων, κυρίω για θύματα εκμετάλλευση σε ένα κράτο μέλο. Και συνειδητά δεν έκανα διάκριση ανάμεσα στι κατηγορίε θυμάτων, τα θύματα που επιλέγουν να επιστρέψουν στη χώρα του και αυτά, τα θύματα που επαναπροωθούνται. Έχουμε ευθύνη θα πρέπει να τους παράσχουμε τις ε, ε, υπηρεσίες είτε επιστρέφουν και ο θελός είτε επαναπροωθούνται. Για τις ε, υπηρεσίες φύλαξη των σύνορων χρειάζεται καλύτερη κατάρτιση ώστε να εντοπίζονται τα θύματα της εμπορίας των ανθρώπων κυρίως όταν πρόκειται για σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι 28 ήταν οι τροπολογίε που κατέθεσαν για αυτή την έκθεση και Αποφάσισα να μην καταρτήσω συμβαστικές τροπολογίες ε, λόγω των δεδομένων ε, ε, και κατάστα και η ίδια δύο τροπολογίε για το στοχο εκκληρια Κιλετία 5-1 για την εγκατάργηση οποιοδήποτε μορφή βία κατά γυναικών και κοριτσιών στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα και επίση σε σχέση με τη, όλα τα είδη εκμετάλλευση σεξουαλική και άλλη. Ε, ευχαριστώ τους συναδέλφους ε, της Επιτροπής για τις τροπολογίες που κατέθεσαν και σε διάφορες τροπολογίες δεν ε, ρίχνουμε το βάρος ούτε στις εξωτερικές σχέσεις, σε αυτήν την εξωτερική διάσταση της εμπορίας ανθρώπων, ούτε στη διάσταση των δύο φίλων. Και όπως και στην Τρουά θα ήθελα και εγώ να διατηρήσουμε την έμφαση σε αυτά τα σημεία και έχουμε και την ξεχωριστή αρμοδιότητα από την Επιτροπή Λίμπε και θα υιοθετήσω την προσέγγιση της κυρίας Λόχ πύλε, ούτως ώστε να ε, προσδοθεί ιδέουσα σημασία στη διάσταση των φίλων κατά την αντιμετώπιση του φαινομένου σε εξωτερικές σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ του αδέλφου που εργάστηκαν πολύ σκληρά μέσα και από τις δικές τους εκθέσεις και προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας. Να περάσω τότε στην ε, έκθεση για την εφαρμογή για την εφαρμογή της οδηγίας. Και πάλι θα ήθελα πάλι να, να ευχαριστήσω τη γραμματεία, τους υπαλλήλους επιτροπής, τους βουλευτές, τις, ε, τους βοηθούς τους και ούτω καθεξής. Για να μην πολυλογώ. 241 ε, θα ήταν οι τροπολογίες ε, και σε βοήθεια, με τη βοήθεια των σκιωδών ε, και των υπαλλήλων καταλήξαμε σε 18 συμβαστικές τροπολογίες που έτυχαν διακομματικής υποστηρίξης κυρίως για τα βασικά στιγμή και τις βασικές παραγράφους της έκθεσης. Θα ήθελα να σας βοηθήσω για τη σύνταξη αυτών των 18 συμβαστικών τροπολογιών. Επίσης, με τους συναδέλφους ε, από ε, την ε, από το ΑΛΔΕ, από τους φιλελεύθερους και από τη διακομματική ομάδα εργασίας για τους ΛΟΑΔΜ καταθέσαμε άλλες τροπολογίες που προσθέτουν κάποια ζητήματα ε, σε σχέση και με τον περιορισμό των αριθμών των χαρακτήρων που μας ε, εμποδίζει από το να συμπεριλαμβάνουμε όλα τα ζητήματα που θέλουμε και επίσης ε, επειδή είναι μεικτή αρμοδιότητα στο ζήτημα και ευχαριστώ παρεμπιπτόντως και τη Μάλιν Μπιόρκ για τη βοήθειά της δεν μπορώ να δεχτώ τροπολογίες που σχετίζονται με αποκλειστική αρμοδιότητα άλλης επιτροπής και ανέφερα ότι αυτές οι τροπολογίες θα πρέπει ενδεχομένω να προσθεθούν στον κατάλογο ψηφοφοριών. Δεν είναι ότι δεν είναι σύμφωνο με τι τροπολογίε, αλλά δεν είναι τη δική μα αρμοδιότητα. Η Επιτροπή ΛΥΒΕ πριν από δύο εβδομάδες ε, έκανε ψηφοφορία για την εξαιρετική τη έκθεση και προσπάθησε να σωματώσει τις, κάποιε απόψει στις δικές τροπολογίε τροπολογίες όπου υπήρχε σύμπνοια με τη δική μα Επιτροπή, κυρίω για το ζήτημα τη πορνεία. Όταν αρχίσαμε να συζητούμε το θέμα, προσπαθήσαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι ε, υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στην ε, εκπόρνευση και στην εμπορία ανθρώπων. Μπορεί να ξαφνιάσει αυτό ε, κάποιους αλλά θέλω να εστιάσουμε την προσοχή μας στο ένα το φαινόμενο, δηλαδή στην εμπορία των ανθρώπων και όχι στην πορνεία αυτή καθ' αυτή ευχαριστώ και πάλι του συναδέλφου για την καταπληκτική συνεργασία που είχαμε και τις τροπολογίες που στόχο έχουν να βελτιώσουν το κείμενο. Ελπίζω να ε, στεφθεί και με επιτυχία, ε, ε, στεφθούν με επιτυχία και οι δύο εκθέσει αύριο στην ψηφοφορία. Τέλεια, ευχαριστώ τη συνάδελφο για την παρουσίαση της. Θα ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Ε, Hvala vam ε, lijepo gospođo ε, predsjednice, zahvaljujem Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η έκθεση και θα ήθελα απλά να σας πω όπως έχω υποβάλει με τους συναδέλφους κάποιες τροπολογίες και αφορούν το θέμα των παρένθετων γονέων. Ελπίζω λοιπόν να τις λάβετε υπόψη, γιατί κάθε χώρα στον κόσμο έχει πολύ αυστηρές ρυθμίσεις ε, για την ε, διακίνηση ανθρώπων ε, και δεν θα πρέπει να υπάρχει κάποια διάκριση για τους παρένθετους γονείς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε το σώμα μιας γυναίκας, το οποίο είναι αντικείμενο εμπορίου και θεωρώ πως αυτό υποβαθμίζει την αξιοπρέπεια των γυναικών. Η πρακτική αυτή η οποία περιλαμβάνει αναπαραγωγική εκμετάλλευση και την χρήση του ανθρώπινου σώματος για χρηματικό όφελος πρέπει να απαγορευτεί. Και αυτό πρέπει να το δούμε στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν δείτε τις διατάξεις ε, της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρεται ξεκάθαρα πως τα συμβαλόμενα μέρη πρέπει να αναλάβουν μέτρα τα οποία σκοπεύουν να προλάβουν οποιοδήποτε είδους εμπορία παιδιών. Και θεωρώ πως η ε, παρένθετη γονείς είναι μια τέτοια περίπτωση. Επίσης υπάρχει μια επιτροπή η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων η οποία καταψήφισε την δυνατότητα αυτή στην Ευρώπη. Οπότε είναι σαφές πως η κοινή γνώμη είναι κατά του θέματος αυτού. Αν δούμε το τι γίνεται και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, νομίζω πως είναι ομόφωνη η στάση, πως πρέπει να απαγορευτεί αυτή η πρακτική και οι πολιτικές ομάδες ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περισσότερες δηλαδή, συμφωνούν. Και οι διάφορες ΜΚΟ που ασχολούνται με τα δικαιώματα των γυναικών. Επίσης, να ευστηθεί την προσοχή σας σε κάτι άλλο. Ο τουρισμός για παρένθετες μητέρες ε, στην Ινδία και στις ΗΠΑ βρίσκεται σε πλήρη άνθηση. Και απέχουμε πάρα πολύ λίγο από το να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέπουμε πως υπάρχει αύξηση της πρακτικής αυτής ε, τα τελευταία χρόνια και θεωρώ πως αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί θα καταλήξει στο να μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους ε, σαν εμπορεύματα. Γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την εισηγήτρια να εξετάσει τις ε, τροπολογίες για την απαγόρευση κυρία Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Οπωσδήποτε πολλή δουλειά έχει γίνει για αυτές τις δύο εκθέσεις και νομίζω ότι καταλήξαμε με συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες γίνονται αποδεκτές από όλες τις πολιτικές ομάδες. Νομίζω ότι είναι επίτευγμα αυτό δεδομένου του αντικειμένου. Ελπίζω λοιπόν να στηρίξουν όλες οι ομάδες τις συμβαστικές προτάσεις και την έκθεση. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω το θέμα αυτό της μείωσης της συζήτηση για την πορνεία. Συμφωνώ με την κυρία Μπίρντερ ότι δεν πρέπει να μπλέκουμε την εμπορία ανθρώπων με την πορνεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, η πλειοψηφία των διακινούμενων ε, σχεδόν όλες. Γι' αυτό το σκοπό διακινούνται. Οπότε η πορνεία είναι μεγάλο κομμάτι του θέματος. Ξέρω πως υπάρχουν και άλλες μορφές διακίνησης ανθρώπων, εξίσου σημαντικές, και καλύπτουν οι εκθέσεις και τις δύο αυτές περιπτώσεις. Η πορνεία είναι μεγάλο κομμάτι των όσων λέμε. και ιδιαίτερα θα ήθελα να επενέσω την τροπολογία 13 στην σελίδα 14 που μιλάει για τη μείωση της ζήτησης. Και νομίζω όλοι στην Επιτροπή μας θεωρούν ότι πρέπει να μειώσουμε την ζήτηση Ε, και θα πρέπει ακριβώς να δούμε τη σχέση, την πιθανή μεταξύ της ζήτησης σεξουαλικών υπηρεσιών και διακίνησης ε, ανθρωπίνων όντων. Και η τροπολογία αυτή θεωρεί πως η μείωση της ζήτησης μπορεί να επιτευχθεί μέσω νομοθεσίας η οποία θα μεταφέρει το βάρος ε, στους πελάτες, σε αυτούς που αγοράζουν τέτοιες υπηρεσίες και όχι σε αυτούς που τις πουλούν. Τα μέλη της Επιτροπής τα οποία είναι εδώ πέρα καιρό θα θυμούνται πως ε, την ε, προηγούμενη Δευτέρα περάσαμε μια έκθεση η οποία λέγε ακριβώς αυτό ότι δεν πρέπει να ποινικο... ότι θα πρέπει να ποινικοποιούμε τον αγοραστή και όχι το θύμα και το ενισχύουμε νομίζω αυτό εδώ και είναι ένα σημαντικό κομμάτι του τι προσπαθούμε να κάνουμε στην έκθεση αυτή και είναι και στην οδηγία την ίδια Αφορά δηλαδή η δεύτερη έκθεση την εφαρμογή της οδηγίας και η μείωση της ζήτησης υπάρχει στην οδηγία, οπότε είναι σημαντικό να το ενισχύσουμε αυτό. Να σας ευχαριστήσω όλους, ε, όλες τις σκιώδεις ηγήτρες και ελπίζω η έκθεση να περάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπιόρκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την Καθρίν Πίρντερ και τις ε, σκιώδεις ε, εισηγήτρες, υπόλοιπες δηλαδή. Εγώ είμαι σκιώδης εδώ στην Επιτροπή και στην ε, Επιτροπή και είμαι και συντάκτρια της έκθεσης στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Θα ήθελα λοιπόν να καταθέσω κάποιες σκέψεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για το περιεχόμενο της έκθεσης, διότι πέρα από τις αρμοδιότητες Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ε, γιατί μην ξεχνάμε ότι περιγράψαν πολύ σωστά τα δικαιώματα των γυναικών χάρη στη ΛΥΜΠΕ και δόθηκε η σημασία στη διάσταση των δύο φύλων, ε, ε, και επίσης ασχοληθήκαμε και με τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ έτσι είμαι ικανοποιημένη για... από το περιεχόμενο και των δύο εκθέσεων και ελπίζω να έχουμε αύριο καλά αποτελέσματα. Στην ε, ψηφοφορία και βλέπουμε πως από πλευράς ε, δικαιωμάτων ο στόχος και των δύο επιτροπών είναι να παρασχεθεί επαρκής προστασία στα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στην έκθεση ασχολούμαστε ενδεχομένως λίγο περισσότερο με τα δικαιώματα ε, των παιδιών και ε, τα, με τα θέματα συνεργασία ε, με τις ΕΠΟΛ, τη Europol, τη Eurojust, όλα τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα δηλαδή που πλαμβάνονται αυτών των ζητημάτων επίσης. Μιλάμε και για το δικαίωμα δικαστική συνδρομής, γιατί αυτό είναι αρμοδιότητα τη ΛΥΜΠΕ και ελπίζω να δοθεί η απαιτούμενη σημασία για αυτό το ζήτημα και στην Επιτροπή Γυναικών. Δηλαδή θα πρέπει να τιμωρούνται τα θύματα ε, για διοικητικές παραβιάσεις ε, που γίνονται όταν κάποιος πέφτει θύμα ενός ε, τέτοιου εγκλήματος και θα πρέπει λοιπόν να παράσχεται η απαιτούμενη δικαστική συνδρομή στα θύματα αυτών των πράξεων. Επίσης, και στις δύο εκθέσεις, όπως είπε και η συνάδελφος Χόρνμελ, είναι σημαντικό να μιλήσουμε για το, το θέμα της καταπολέμησης της ζήτησης. Δεν μιλάμε για την πορνεία, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να τολμήσουμε να αποδώσουμε τις ευθύνες, ε, κυρίως διότι συνδέονται τα δύο ζητήματα. Και Βαρέθηκα να διαβάζω ότι πρέπει να καταρτήσουμε τις γυναίκες και ότι πρέπει να μάθουν τα κορίτσια και τα γυναίκες να αντιμετωπίζουν αυτά τα ζητήματα. Κουράστηκα με αυτή την προσέγγιση και νομίζω ότι θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας στους άντρες. Ε, πώς θα τους κάνουμε να σταματήσουν σταματήσουν να αγοράζουν ε, σεξουαλικές υπηρεσίες. Ε, νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα πραγματικό βήμα για να έχουμε μεγαλύτερη ισότητα και για να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικότερα το φαινόμενο της πορνείας και ε, άρα και της εμπορίας ανθρώπων. Εάν περάσουν αυτά που προτείνει η Επιτροπή Ελευθεριών, πώς να το πω στα Σουηδικά, Ε, όποιος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ενός θύματος εμπορίας ανθρώπων, εκείνου η πράξη θα πρέπει να ποινικοποιείται. Ε, δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή περιγραφή αξιόπινης πράξης, αλλά έχουμε καταλήξει σε ένα μέτρο, σε μια συμβαστική τροπολογία μέσα στην έκθεση της Επιτροπής Ελευθερίων και λέμε ότι όποιος συνειδητά χρησιμοποιεί αυτές τις υπηρεσίες ε, του θύματος ε, της εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει ε, αυτόν η πράξη να ποινικοποιείται και νομίζω ότι είναι ικανοποιητική αυτή η διατύπωση με τις ε, τροπολογίες που έχουμε καταθέσει. Ενισχύουμε την διοικητική και τη δικαστική συνεργασία για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου και ήταν πολύ καλή συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μπιόρκ. Τώρα, Δόκτωρ Γκάρετ Ομπράιν από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μας καλέσατε σήμερα εδώ για να σχολιάσουμε αυτή την τόσο σημαντική γνωμοδότηση της Επιτροπής σας. Καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον της Επιτροπής σας ε, για το θέμα αυτό. Εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την εμπορία ανθρώπων στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουμε με τρίτες χώρες ως θέμα που άπτεται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του φύλου. Η διακίνηση ανθρώπων ε, αντιμετωπίζεται και σε άλλους διαλόγους πολιτικής ε, με τρίτες χώρες. Ενθαρρύνουμε συνεχώς ε, τις τρίτες χώρες να αντιμετωπίζουν την ε, εμπορία ανθρώπων ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και να υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση και να υπάρχει κατάλληλη υποστήριξη για τα θύματα. Είχαμε και κάποιες πρόσφατες εξελίξεις στην εξωτερική διάσταση. Το 2015 είχαμε το νέο πρόγραμμα δράσης ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία έδωσε προτεραιότητα στην εμπορία ανθρώπων και έδωσε προτεραιότητα και στα δικαιώματα των προσφύγων που είναι ε, θύματα εμπορίας ε, και θέλουν να βοηθήσουν και την κινητικότητα και διάλογο με τρίτες χώρες και την κύρωση και εφαρμογή κομβικών ε, διεθνών συμβάσεων για θέματα εμπορία ανθρώπων. Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί προτεραιότητα και στο πλαίσιο των ε, δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ισότητα ε, των Φύλων και για την αντινόμηση των σχέσεων το 2016-2020 για να ε, καταπολεμάται η εμπορία γυναικών και κοριτσιών για όλες τις μορφές ε, ε, θυμάτων και επίσης θέλουμε να παράσχουμε βοήθεια στις γυναίκες που είναι θύματα εμπορίας, κυρίως ε, τις οβάλλοντες ομάδες, Γι' αυτό ακριβώς και συνεχίζουμε να θεωρούμε προτεραιότητα την εμπορία ανθρώπων σε θέματα μετανάστευση και εξακολουθούμε να το τηρούμε αυτό και κατά την πορεία μας προς μια νέα στρατηγική για την εμπορία ανθρώπων σε στενή συνεργασία με τους ε, ε, συναδέλφους που είναι ε, στη Γενική Διεύθυνση HOME στο Τμήμα Καταπολέμησης της εμπορία Ανθρώπων. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριο Μπράιαν. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια για τα τελικά συμπεράματα. Μετά, κυρία Μπίρτερ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Κάποια πράγματα θα ήθελα να φέρω. Οι γονείς είναι δύσκολο θέμα. Γιατί αντιμετωπίζουν διαφορετικά οι χώρες. Σε κάποιες χώρες επιτρέπεται, σε άλλες όχι. Σε άλλες επιτρέπεται η πληρωμή, σε άλλες όχι. Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες ε, για την δωρεά οαρίων ε, και, τον, και τις διάφορες πρακτικές και είναι δύσκολο να το απογνώσουμε και οι τροπολογίες δεν ήταν στις συμβαστικές προτάσεις και θα ψηφιστούν χωριστά. Αλλά όσον αφορά την διακίνηση προσώπων νομίζω πως ε, η παρένθετη γονείς δεν είναι ένα τέτοιο θέμα το τι συμβαίνει μετά στα βρέφη και η καταναγκαστική φύση ε, άλλων περιπτώσεων ε, βεβαίως είναι πολύ δύσκολα ζητήματα. Οπότε οι τροπολογίες σας θα ψηφιστούν χωριστά αύριο. Μείωση της ζήτησης, ναι, συμφωνώ. Οποιαδήποτε διακίνηση υπάρχει γιατί υπάρχει ζήτηση και ξέρουμε πως τεράστια πλειοψηφία των θυμάτων είναι γυναίκες που πάνε στον κλάδο του αγοραίου έρωτα. Και πώς θα μειωθεί η ζήτηση ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά οι τροπολογίες που ασχολούνται αποκλειστικά με την πορνεία είναι ελαφρώς διαφορετικές. Κάποιες μπήκαν στις τροπολογίες, κάποιες όχι. Οι υπόλοιπες θα ψηφιστούν ξεχωριστά. Ευχαριστώ και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και το γεγονός ότι για τα λόγια που είπατε και για το γεγονός ότι πλέον θα θίγεται αυτό το ζήτημα. Αλλά έχουμε και το ζήτημα της επιστροφής των θυμάτων που έχουν υποστεί κάποια τραύματα ψυχολογικά. Όποια και αν ήταν η μορφή της διακίνησης. Δηλαδή καμιά φορά φεύγουν ε, πιστεύοντας ότι πηγαίνουν κάπου καλύτερα και λένε στην οικογένειά τους ότι ε, για αυτό πάνε. Και μετά όταν επιστρέφουν χρειάζονται και κάποια ιδιαίτερη φροντίδα. Γιατί υπήρχαν βεβαίως και οι προσδοκίες που διαψεύστηκαν. Και κυρώσεις που υφίστανται για τη δουλειά που εξαναγκάστηκαν να κάνουν. Σας ευχαριστώ λοιπόν και περιμένω το σχολείο σας αύριο. Ευχαριστώ κυρία Μπίρντερ. Όπως ε, πολύ σωστά είπε και η συνάδελφος, αύριο θα γίνει η ψηφοφορία αυτών των δύο εκθέσεων. Περνάμε τώρα στο σημείο 6 γνωμοδότηση για την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, η συμβολή του Κοινοβουλίου εν ώψη της πρότασης της Επιτροπής. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης είναι η κυρία Μούτη, η οποία όμως δεν είναι εδώ. Δεν μπορούμε λοιπόν να συζητήσουμε την έκθεση αυτή γιατί λείπει η συντάκτρια να σας ε, υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ε, για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση είναι 25 Απριλίου στις 5 και θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση στις 24 Μαΐου στη συνεδρίαση της Επιτροπής Γυναικών. Λύεται συνεδρίαση. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 10 μετά από τις συνεδρίες των συντονιστών για τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ.